Σα ευχαριστώ. Συνάδελφοι, προσέξτε, θα πρότεινα να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τους Ευρωπαίους Χριστιανοδημοκράτες και την ομάδα των Πρασίνων, την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, τις εξής προτάσεις, τους εξής διορισμούς, διορισμούς με συγχωρείτε, για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φίλων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ, για την κοινή ε, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κροατίας, η κυρία Κορνέλισεν που θα λάβει την θέση της κυρία Χάιντερ Ρούλε. Υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Αυτοί οι διορισμοί λοιπόν επικυρώνονται από το σώμα. Sorry. Point of order. Συγγνώμη, διαδικαστικό εσείς. Yes, okay. Παρακαλώ. Uh, Κοιτάξτε, επειδή ο σεισμός στην Ιαπωνία και η καταστροφή στην Ιαπωνία συνέβησαν πρόσφατα, ήταν δεδειγμένο το Κοινοβούλιο μαζί να υποστηρίξει το λαό της Ιαπωνίας τη Δημοκρατία τη Ιαπωνία εκφράζοντα συλληπιτήρια και τηρώντα ενό λεπτού σιγή για τα θύματα τη Ιαπωνία. Προσέξτε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνεδρίαση όλων των Ευρωβουλευτών